Καλωσορίζω για μια ακόμη φορά την κυρία Αντιπρόεδρο, την υπάτη εκπρόσωπο. Υπάρχει επίσης εκπρόσωπος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα είναι η εταιρική σχέση με την Ανατολική Ευρώπη, η Ανατολική εταιρική σχέση και η συνάντηση κορυφής που θα οργανωθεί στη Βαρσοβία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Κύριε Πρόεδρε, λέει δηλαδή Άστον, είναι μεγάλη χαρά για μένα που απευθύνομαι σε εσά πριν από τη συνάντηση κορυφής ε, που θα γίνει στη Βαρσοβία 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε συστηματικά την εταιρική ανατολική σχέση και εσείς Πρόεδρε θα πάρετε το λόγο εξ του Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω και εσάς πρόεδρε και τον Στέφεν Φούλε, ο οποίος έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για την ανατολική εταιρική σχέση. Η ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεών μας με τους γείτονές μας είναι βασική προτεραιότητα και θεωρώ ότι είναι η βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια προτεραιότητα από την οποία θα κρυθούμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στους ανατολικούς μας γείτονες τα τελευταία 20 χρόνια εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε τη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μόνο προς το δικό σου συμφέρον αλλά και το δικό μας, γιατί βελτιώνει και τη δική μας ασφάλεια και ευημερία. Τον Μάιο του 9 ξεκινήσαμε την Ανατολική Εταιρική Σχέση σαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα οικοδομήσουμε την πολιτική μας σύνδεση και την οικονομική μας ολοκλήρωση με έξι χώρες, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Κάναμε βήματα προόδου τα τελευταία δύο χρόνια, ενισχύσαμε τις διμερείς μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Φέτος θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία και στα πλαίσια της ε, σε βάθος ε, συνολικής ζώνης ελευθέρου εμπορίου. Επίσης έχουμε προχωρήσει ε, προς την κατεύθυνση αυτή και με τη Γεωργία και την Μολδαβία. Επιπλέον έχουμε κάνει βήματα και στον τομέα της κινητικότητας των πολιτών. Εφαρμόζουμε προγράμματα δράσης για θεωρήσεις με Ουκρανία και Μολδαβία και συμφωνίες επανεισδοχής με την Γεωργία εδώ και λίγους μήνες. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις και με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία στο μέλλον. Στη Βαρσοβία θα συναντηθούμε στα πλαίσια αυτών των στενών σχέσεων λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν ενώνει μόνο κυβερνήσεις αλλά λαούς. Υποστηρίζω τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους ομολόγους του στην Ανατολική Ευρώπη μέσω της Euronest, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest. Η κοινωνία των πολιτών και τα επιχειρηματικά φόρουμ έχουν συνέλθει στα πλαίσια αυτής της εταιρικής σχέσης και πήρε μέρος ο Στέφεν Φούλε. Πέραν αυτού, τα τελευταία τέσσερα χρόνια άνω των 2.000 φοιτητών και καθηγητών πανεπιστημίου από χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση ε, ήρθαν χρηματοδοτούμενοι να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα ε, προχωρήσουμε στην υπευθυνοποίησή μας, στην αμοιβαία υπευθυνοποίηση και σεβασμό των αρχών της δημοκρατία, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Νομίζω ότι έτσι θα προωθήσουμε και τις ευρωπαϊκές επιλογές και τις ευρωπαϊκές προσδοκίες έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν σε μια δημοκρατία βιώσιμη και υποστηρίξιμη. Πράγματι έχουμε τύχει υποστήριξης από τους εταίρους μας στην προσπάθεια αυτή Εγώ μετέφερα το θέμα αυτό στην Ουκρανία πρόσφατα, λέγοντας ότι οι δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, όπως και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, είναι βασικές αρχές και βάση των σχέσεών μας. Ο Στέφεν Φούλε και εγώ ανησυχούμε για την διαδικασία τη δικαστική εις βάρος της Γιούλια Τιμοσένκο και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Όπως ήδη είπα, ο Στέφεν Φούλε συνεργάζεται με τους Ουκρανούς τον τελευταίο καιρό, μεταφέρει τα μηνύματά μας και αναπτύσσει μια τέτοια σχέση σε βάθος για να προχωρήσουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς ε, είμαστε επίσης ξεκάθαροι σε σχέση με την κατάσταση ε, της καταπίεσης των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και στις τελευταίες εκλογές. Επιβάλαμε μετά τις εκλογές κυρώσεις εις βάρος του καθεστώτος και ζητήσαμε να απελευθερωθούν και να αποκατασταθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ταυτόχρονα αυξήσαμε τη βοήθειά μας προς την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Μετά από την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας, την οποία ξεκίνησα και εγώ και ο Φούλε, νομίζω ότι θα επιβάλλουμε ακόμα περισσότερες προϋποθέσεις στα πλαίσια των δράσεων της πολιτικής αυτής γειτονίας. Αυτό σημαίνει περισσότερη οικονομική στήριξη, στενότερη πολιτική συνεργασία, βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση με όλους αυτούς τους εταίρους που έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις σε βάθος. Όλο και περισσότερο, για όλα και περισσότερο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη διάσταση θα μας επιτρέψει να στρέψουμε ένα τμήμα της βοήθειας και προς μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό με το μέσο στήριξης της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Γειτονίας. Θα υποστηρίξουμε έτσι λοιπόν και το μέσο για τη δημοκρατία ε, στην περιοχή αυτή. Και ευχαριστώ όλους όσους μας συμβουλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι συγκρούσεις στην περιοχή, στο Άνω Καραμπάχ, στην Υπερνιστερία, την Αμπχαζία και, ε, και την Νότια Οσετία είναι τα ανησυχητικά εμπόδια ε, μπροστά στα βήματα πρόοδο που πρέπει να γίνουν. Περιμένουμε λοιπόν από τους ανατολικούς εταίρους να κάνουν προσπάθειες όπως και εμείς κάνουμε προσπάθειες στα πλαίσια αυτής της περίπλοκης σχέσης. Τον Αύγουστο μετά από σύστασή μου το Συμβούλιο ενέκρινε το διορισμό του Φιλίπ Λεφόρ τον, σαν, στον διορισμό του Φιλίπ Λεφόρ σαν ειδικό ε, ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάυκασο και την κρίση στη Γεωργία σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και συνεργαζόμενοι στενά με όλους τους εμπλεκομένους. Το Άνω Καραμπάκ παραμένει πράγματι ψηλά στην πολιτική μα ατζέντα. υποστηρίζοντα τη διαδικασία τη ομάδα του Μίνσκ είμαστε σε διάλογο με όλε τι πλευρέ. Έχουμε την επιθυμία και την ικανότητα να αναλάβουμε δράση υπέρ κάποιων προσπαθειών αποκατάσταση και σταθεροποίηση τη σύγκρουση. Όπω ακριβώ το δείξαμε και μετά τον πόλεμο στη Γεωργία. Στην υπευνηστερία η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε το ρόλο της που οδήγησε στην απόφαση για την εκκίνηση των νέων διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Φόρμουλα 5 2. Η απόφαση ελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τώρα με καλή θέληση και καλή την πίστη θα προχωρήσουμε σε συνεργασία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να δώσουμε μια νέα όφηση στην δημιουργία στενών σχέσεων με τους ανατολικούς μας εταίρους και γείτονες και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η δημοκρατία και να επικρατήσει το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο συνάδελφος Έλμαρ Μπρόκ από το ΕΛΚΑ έχει τώρα το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλώ κυρία Άστον, κύριε Επίτροπε. Γιατί μιλάει για το Συμβούλιο η κυρία ε, Άστον, ε, δηλαδή γιατί κάθεται στα έδρανα του Συμβουλίου, γιατί είναι κοινοτική η πολιτική, πρέπει να είναι στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά μπορεί να μου απαντήσει. Ε, ελπίζω η Σύνοδος Κορυφής στη ε, Βαρσοβία να στεφθεί με επιτυχία και παρά τις διαφορετικές εξελίξεις στις διαφορετικές χώρες πρέπει να τονίσουμε εδώ τη Λευκορωσία, ε, ελπίζουμε να πετύχουμε την πολυμερή ε, συνεργασία. Ε, υπάρχουν υπαγωμένε σειράξει σειράξεις παράδειγμα το ορεινό Καραμπάχ, θα μπορούσε να λύσει κανείς πιο εύκολα τέτοιες διενέξεις αν συνεργαζόντουσαν περισσότερες χώρες μεταξύ τους γιατί έχουν και κοινά συμφέροντα και για οικονομικούς και για πολιτικούς λόγους θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η πολυμερής προσέγγιση στην εταιρική σχέση για να προχωρήσουμε και στα οικονομικά αλλά και στα πολιτικά θέματα. Είναι σημαντικό σε χώρε όπως η Λευκορωσία να τονίσουμε ότι ε, θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τα κόμματα της ε, αντιπολίτευσης και τη κοινωνία των πολιτών εφόσον δεν υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Να χρησιμοποιήσουμε τις δομές για να παρακάμψουμε την κρατική μηχανή και να προωθήσουμε τα αιτήματα για τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Κυρία Άστον και κύριε Φούλε, επιτρέψτε μου και μια ακόμα παρατήρηση που έχει να κάνει με τα σημερινά γεγονότα. Άκουσα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας στην Ουκρανία σήμερα βάσει ενός άρθρου του ποινικού κώδικα που είναι εμπνεύσεως του Στάλιν από το 1957 και το 1962 ενισχύθηκε λίγο ζήτησε 7 χρόνια φυλάκιση κατά της κυρίας Τιμοσέγκο με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Και επίσης θα πρέπει να διαπιστώσουμε περαιτέρω ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση Τιμοσέγκο, αλλά είναι 15-16 εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς. Αν μέχρι την Παρασκευή δεν υπάρξει καμία δήλωση και ε, θα πρέπει να, δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Συζητήσαμε με τον κύριο Μπίλτ, με τον κύριο Φίλε για το τι θα κάνουμε απέναντι στον κύριο ε, Κόβιτς γιατί ε, είναι και προς το συμφέρον μας να γίνει η συμφωνία με την Ουκρανία αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μια χώρα που θέλει να έχει και ευρωπαϊκή προοπτική θα πρέπει να τηρεί τα στοιχειώδη της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος Χάνες Σφόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κυρία Άστον για την προσήλωσή σας στη ε, γειτονία και για τον κύριο Φίλε, ο οποίος κάνει πάρα πολύ εντατικέ προσπάθειες, όχι μόνο για τη σχέση γειτονίας αυτή καθ' αυτή, αλλά και για τον εκδημοκρατισμό των κρατών. Ε, επιτρέψτε μου να πω ευθύ εξ αρχή ότι αυτό που μα ενδιαφέρει στην ανατολική εταιρική σχέση δεν είναι να συμμαχίσουμε απέναντι στη Ρωσία. Όχι, να συμμαχίσουν μεταξύ οι χώρε αυτέ, Είναι ελεύθερη τους ε, βούληση και απόφαση προ τα που θέλουν να προσανατολιστούν και αν θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Ρωσία ενδεχομένω σε άλλο είδο συνεργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ουκρανία. Για μας είναι πολύ σημαντικός εταίρος και εύχομαι κάθε επιτυχία στη διάσκεψη στην Πολωνική Προεδρία. Γνωρίζουμε ότι έχει σχέση και με την κατάσταση στην Ουκρανία. Και πρέπει να πω το εξή. Ο πληθυσμό αναρωτιέται στην Ουκρανία και δικαίω. Πώ προέκυψε αυτή η συμφωνία με τη Ρωσία για τι τιμέ του φυσικού αερίου, Πώ ξαφνικά έγινε από εχθρό τη Μοσέγκο η Ρωσία φίλο τη, που την υπερασπίζεται κιόλα. Εξ όσων γνωρίζω, η τιμή αυτή που συμφωνήθηκε δεν είναι και πάρα πολύ ευνοϊκή για το λαό της Ουκρανίας. Μπορεί να θεωρηθεί μέχρι και αρνητική. Πάντως είναι σαφέστατη η θέση και της δικής μου πολιτικής ομάδας. Αυτά τα θέματα λύνονται και αντιμετωπίζονται πολιτικά και όχι με ποινικά δικαστήρια. Γι' αυτό απευθύνουμε και έκκληση σαφή και στον Πρόεδρο και στην κυβέρνηση της χώρας να βρει ε, μία διέξοδο από την κατάσταση που έχει προκύψει. Η καταδίκη της κυρίας Τιμοσέγκο Νομίζω τότε που είπες ε, ε, Μπρόκ για τον Στάλιν είχε ήδη πεθάνει, είπε στο 57. Εν πάση περιπτώσει, είχε αποβιώσει τότε ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία. Όπως και να έχει η νομική ε, κατάσταση και η ένομη τάξη στη χώρα, είναι απαράδεκτο με πολιτικούς σκοπούς να διώκεται κάποιος ποινικά στα δικαστήρια. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πατή Εκπρόσωπο και το Κοινοβούλιο να διατρανώσει ότι θέλουμε να έχουμε κοντά μα ε, την Ουκρανία, μια δημοκρατική Ουκρανία με πολιτικού ε, στόχου που να του επιδιώκει όμω με πολιτικά μέσα. Ελπίζω να το καταλάβουν και να ε, πάρουν και αυτό το δρόμο για την αλλαγή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Έχετε απόλυτο δίκιο και οι δύο συνάδελφοι που αναφέρεστε στον Επίτροπο Φίλε. Σα ευχαριστώ που είστε μαζί μα κατά τη διάρκεια τη είναι πολύ κοντινοί μας γείτονες. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γκέρμπερ Γιάνν Γεμπράντι, εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρία είπατε εκπρόσωποι. Ε, είναι γνωστό ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Είναι αμοιβαία η συνεργασία. Το λέμε και ε, σε άλλες περιοχές και στην Αφρική και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή και μοιραζόμαστε την ίδια πίστα χορού και στροβελιζόμαστε μάλιστα. Ενώ ε, στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Εκτός από τη Σουηδία και την Πολωνία δεν ενδιαφέρονται οι πολίτες ούτε οι χώρες να τονωθούν οι σχέσεις μας και να ενισχυθούν με την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι κοντόφθαλμο. Γιατί έχουμε συμφέρον να είναι οι γειτονέ μας σταθεροί ε, για να είμαστε και εμεί σταθεροί, αρκεί και μόνο να αναφέρουμε την εξάρτησή μα για θέματα ενέργεια από την περιοχή. Και θέλω να ρωτήσω και την Επίτροπο, την κυρία Άστον και τον κύριο Φίλε, τι θα κάνουν για να λάβουν πρωτοβουλία για να εμβαθυνθεί ο πολιτικός ε, διάλογος. Να μην είναι χωροδιδάσκαλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρτενέρ του χώρου θα πρέπει και στην ε, ε, Ουκρανία να δούμε τη γίνεται και ανησυχώ πολύ και για το Ζαρμπαϊτζάν και για τη Λευκορωσία που συλλαμβάνονται οι αντιφρονούντες. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε και σε αυτή την πίστα και να χορέψουμε και στην Ανατολική Ευρώπη, να είναι πιο εύκολα τα ταξίδια και για μας και για τους εταίρους μας εκεί. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν όροι και ε, προϋποθέσεις, αλλά το να στρέφουμε την πλάτη ο ένας στον άλλον δεν βοηθάει. Ευχαριστώ την κυρία ε, Άστον ε, για ε, τη συνεργασία που έχει με δημοκρατικές δυνάμεις όπως είναι και στο Αζερβαϊτζάν. Εκτός από τη Ρωσία μπαίνει στο χορό και η Τουρκία τώρα. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι ένα όραμα και μια προσήλωση. Πριν από δύο χρόνια για πρώτη φορά συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο με τους πέντε της Euronest. Η Λευκορωσία δεν είχε προσκληθεί τότε ούτε καταλήξαμε σε μια κοινή δήλωση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω στη διαδικασία και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούμε ένα τον άλλο να συνεργαζόμαστε για να βγει κάτι όμορφο στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Συνάδελφος ε, κύριος Τάνοκ, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιάσει στην νότια διάσταση, ε, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, αλλά δεν πρέπει να χάρουμε και τη σημασία των ανατολικών εταίρων μας και την υποστήριξή μας ε, για πιο στενές σχέσεις με τις έξι αυτές χώρες. Η Ουκρανία διέρχεται μια πολύ δύσκολη φάση, υπάρχει επιδείνωση στις δημοκρατικές της δομές, στο κράτος δικαίου, όπως ε, διαπιστώσαμε με την επιλεκτική δικαιοσύνη που εφαρμόστηκε στην Γιούλια Τιμοσέγκο η Λευκορωσία εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια ενός δικτάτορα του Λουκασέγκου. Και η κατάσταση στον Κάφκασο είναι ανησυχητική γιατί η Ρωσία εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή της ε, τη Γεωργία αυξανόμενη ένταση στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία για τον Αγκόρνο Καραμπάχα. Ε, χαίρομαι που ορίστηκε ε, εντεταλμένος για την περιοχή αυτή πριν από δύο εβδομάδες στη Euronest το αδιέξοδο με βάση το άρθρο για τις τρίτες χώρες ε, περιλαμβάνει και τις ε, τρεις δημοκρατίες ε, του Καυκάσου και πλέον έχουν παραλύσει οι διαδικασίες, δεν προχωράνε καλά για τη συνεργασία με τη Euronest. Ελπίζω λοιπόν ότι στη διάσκεψη κορυφή στη Βαρσοβία δεν θα γίνει, δεν θα καταλήξει όπως με αυτό που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εστιάσει την προσοχή της σε πραγματιστικά θέματα όπως είναι η βίζα και η απελευθέρωση του εμπορίου και όχι με άπιαστα τα θέματα. Uh, Ζητώ ε, συγγνώμη από εσάς, ε, δεν σας ε, είχα δει, δεν είχα δει που ήρθατε εδώ στην αίθουσα εκπροσωπώντας στην Πολωνική Προεδρία ο κύριος Βένα Σούλτς από τους Πράσινους Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η νεοσυστασίσα αρχή More for θα πρέπει να ισχύει κυρίως στους ανατολικούς εταίρους μας για την βελτίωση της κοινωνίας των πολιτών που προσφέρει πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου μπορούμε να συνεργαστούμε και με την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ θερμά κυρία Άστον και κυρία Επίτροπε Φίλε να μεριμνήσετε έτσι ώστε το φόρουμ αυτό να αποκτήσει γραμματεία στις Βρυξέλλες και με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί η εργασία του. Γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι κάνουν, ε, το κάνουν ε, εκτός ε, χωρίς αμοιβή και έχουν φτάσει τα ωριά τους. Το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά βλέπουμε και από τις αντιθέσεις που προέκυψαν στη Euronest. Υπάρχουν περιφερειακές συγκρούσεις που παρεμποδίζουν τη συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν η επίλυση των διαφορών θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνεργασία μας με τους εταίρους. Κυρίως στην περίπτωση της υπερδνηστερίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει μόνο ως παρατηρητής στη συζητήση 5 2 και δεν έχει την απαραίτητη εξουσία διαπραγματεύσεων. Στη Βαρσοβία ελπίζω ότι θα επιτύχετε την αποκατάσταση όλων των προσφύγων στη Λευκορωσία και θα καταστήσετε σαφές ότι από εκεί εξαρτώνται πάρα πολλά άλλα πράγματα. Στη τελική ανάλυση πρέπει να συμπεριληφθεί και η Ρωσία στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εύχομαι σε όλους σας καλησπέρα και δίνω τον λόγο στον κύριο Μαστάκα, ε, τον εκπρόσωπο της ΕΓΚΟΕ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ Κάθε βελτίωση των ειρηνικών σχέσεων και της συνεργασίας στην Ευρώπη αξίζει την υποστήριξή μας. Δεν είμαι όμως πολύ βέβαιος για το ποιες είναι οι προθέσεις εκείνων που ε, φύβραν την Ανατολική Γειτονία. Παρ' όλα αυτά ελπίζω η μελλοντική διάσκεψη να βοηθήσει ε, και να μην ε, δημιουργήσει ένα νέο υγειονομικό κλειό και πάλι γύρω από τη Ρωσία. Στη Βαρσοβία θα πρέπει να εκφραστεί η βούληση ότι θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε ε, από την Ιρλανδία μέχρι τα Ουράλια, ενωμένοι στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κατάσταση και να λύσουμε παγωμένες σειράξεις τύπου Ορεινού Καραμπάχ. Θα χαιρόμουν εάν οι διαπραγματευτές στην Ένωση μάθουν να ακούνε και τους συνομιλητές αντί να δείχνουν πάνω αυτή την αλαζονία κάνοντάς του μάθημα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχει το λόγο ο εκπρόσωπος της Ομάδας Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Ήμπρασσας. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η επερχόμενη συνάντηση κορυφής στη Βαρσοβία θα είναι μια καλή ευκαιρία για να διαπιστώσουμε το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και για να βρούμε τις σωστές στρατηγικές γραμμές για αυτή την εταιρική σχέση. Απαιτείται κατά τη διάρκεια αυτής της ε, συνάντησης κορυφής να δοθεί η ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ε, ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και ε, για τις νέες μονάδες. Ξέρετε ότι οι Ρώσοι θέλουν να οικοδομήσουν νέες μονάδες στα ανατολικά μας σύνορα κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα οικολογικά και προβλήματα ασφάλειας όχι μόνο στις χώρες αυτές αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να στρέψουμε την προσοχή μας και στα θέματα διευκόλυνσης ε, της χορήγησης θεωρήσεων. Συμφωνώ με τις προτάσεις του κ. Σβόμποντα για την ανάγκη να υπάρξει επίσης και μία λύση για το περίπλοκο θέμα της Γιούλια Τιμοσέμκο. Άλλωστε θα είναι και μια προτεραιότητα της δικής μου χώρας στην επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε την γυτνίαση της διαδικασίες αυτές ε, ε, στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας και κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μέλτσερ έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στόχος είναι οι έξι πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες να υποστηριχθούν για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ε, και προφανώς η Ρωσία είναι λίγο απορριπτική, το γνωρίζουμε. Η ανατολική σχέση αντιμετωπίζει τις χώρες αυτές ως πιθανά μέλη κάποια στιγμή της Ένωσης. Ε, Συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών έχει προγραμματιστεί με την Ουκρανία και από αυτό θα εξαρτηθεί Εάν θα έχει κάποια δίκαιη δίκη, κυρία Τιμοσέχο, ε, ε, ταυτόχρονα έχουν παγώσει οι ε, διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία. Μια απλή προοπτική της Ένωσης δεν αρκεί για να ενισχύει η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και εσωτερική ειρήνη διαμαγείας. Αυτό φαίνεται και από το παράδειγμα της Τουρκίας και επίσης το τελευταίο δικτάτορα της Ευρώπης, το Λουκασέγκο κάθε φορά που χρειάζεται την Ευρώπη απελευθερώνει ε, που είναι στη φυλακή και πρόσφατα άφησε κάποιους ελεύθερους γιατί έχει τεράστια ανάγκη ε, χρημάτων που δεν βοήθησαν ούτε τα δισεκατομμύρια που τους έδωσε η Κίνα. Για μας όμως σημαντικά κριτήρια αυτά που απορρίπτει ο Λουκασέγκο. πρόεδρος. Και τώρα... Ακολουθούν οι λοιποί ομιλητέ. Ο πρώτος, ο κύριος Χακμάρκ. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Η συνάντηση κορυφή στη Βαρσοβία θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα υποστήριξης και ενημέρωσης επίσης ε, για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε θετικές εξελίξεις στις κοινωνίες αυτές. Όλες οι χώρες αυτές ταλαντεύονται ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, είτε προς απολυταρχικές δομές, είτε προς δημοκρατικές σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι δυνατότητες τις οποίες θα χάσουμε σήμερα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις κερδίσουμε εκ νέου στο μέλλον. Έχει σημασία λοιπόν να τονίσουμε ότι μιλάμε για την Ευρώπη και μιλάμε για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η Ουκρανία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Ιουλία Τιμοσένκο μας το δείχνουν καλύτερα. Η υπονόμευση του κράτους δικαίου είναι μία επιλογή. Από την άλλη είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία ανοιχτή κοινωνία. Έχει πολύ σημασία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία έχει τη διάθεσή της. Είμαστε η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο. Έχουμε τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, ενισχύσεων, επιδοτήσεων και ταυτόχρονα στέλνουμε και ξεκάθαρα μηνύματα για τις προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν εφόσον επιθυμείτε στενότερες μορφές συνεργασίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει στη συνάντηση αυτή κορυφής να δείξουμε ακριβώς τι εννοούμε και τι πρέπει να πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίβετς έχει το λόγο εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πράγματι η ανατολική γειτονία έχει αποδείξει ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και τον αρμόδιο επίτροπο για την εξωτερική ανακοίνωση την οποία έκανε και επιβεβαίωσε το ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση η ανατολική ε, εταιρική σχέση θα πρέπει να βασίζεται σε διαφορετικές πολιτικές γραμμές θα έλεγα για να αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο διαφορετικές χώρες μεταξύ τους όπως η Μολδαβία και το, το Αζερβαϊτζάν. Ζητάμε πολλά, δίνουμε πολλά. Αλλιώς αν δεν δώσουν πολλά δεν θα δώσουμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική μας και αυτό είναι κάτι που θα ενισχύσει τη δημοκρατία γιατί πολλές φορές υπάρχουν αντιλήψεις οι οποίες επικρατούν στις χώρες αυτές που δεν είναι αυτές που περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η Βαρσοβία είναι μία από τις πρωτεύουσε και τις χώρες φυσικά η Πολωνία που προωθούν τις σχέσεις στενής συνεργασίας με την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Η Ουκρανία για μας είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ σημαντική χώρα Γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το δικαστικό σώμα στην ε, Ουκρανία βέβαια, αλλά δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε τις στρατηγικές μας ε, προτάσεις με τα τακτικά μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρουμε. Έχει σημασία να φέρουμε τον κόσμο αυτό κοντά στην Ευρώπη και να επικοινωνούν οι πολίτες των χωρών αυτών ελεύθερα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, εκεί χώρες αυτές για να βοηθήσουμε την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο αγόρευσή σας. Η κυρία Γέτεν Μάκη έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κοινωνία των πολιτών και η πολυφωνία στον πολιτικό πολιτισμό είναι απαραίτητη για όλα τα μέλη μας και όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Γι' αυτό καλωσορίζω την ιδέα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας κοινωνίας των πολιτών που εγκρίνατε στην αναθεώρηση τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, αυτή δεν είναι τελείως ξεκάθαρη για μένα. Άστον. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Άστον, πώς θα αναπτύξει αυτή τη διευκόλυνση της κοινωνίας των πολιτών και ποιος ο ρόλος της στην πολιτική γειτονίας σε σχέση με την τόσο πολυσυζητημένη ιδέα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, European Endowment for Democracy. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Καμίνσκι τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Άστον, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξη για τη γεωργία σήμερα, παραμονές της Συνόδου Κορυφής. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εδαφική ακαιρότητα της γεωργίας είναι ένα θέμα αξιοπρέπειας για τη Δύση. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι επίσης πολύ σημαντικό τμήμα της σημερινής συζήτησης. Παρόλο που Καθόλου δεν θαυμάζω τον πρόεδρο Γιανουκόβιτς, Θέλω να πω ότι δεν θα ήταν σωστό τώρα να συγκρίνουμε την κατάσταση στην Ουκρανία σήμερα με την κατάσταση ε, που επικρατούσε τον καιρό του Στάλιν. Δεν είναι καλή η σύγκριση αυτή και μάλιστα από εκείνου που σιωπούν κατά τα άλλα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Και αν οι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία και καλά κάνουν και τα εκφράζουν, ε, θα περίμενα από εκείνους και τα πολιτικά τους κόμματα να ενδιαφέρονται εξίσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπου ε, κηρύσσονται παράνομα πολιτικά κόμματα, δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές η ε, Βουλή της ε, Ουκρανίας κατά 50% είναι μέλη της αντιπολίτευσης περίπου. Σας ευχαριστώ κύριος Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εταιρική σχέση, η ανατολική εταιρική σχέση έχει μια πολύ σημαντική πολιτική διάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα εμπόδια που αντιμετωπίζει είναι ανησυχητικά. Ο διάλογος με τη Λευκορωσία παραμένει δύσκολος. Ε, στην Ουκρανία η περίπτωση Τιμοσέγκο δείχνει έλλειψη σεβασμού ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεωργία και Αζερβαϊτζάν, ένα κομμάτι του εδάφους του είναι υποστρατιωτική κατεχή κατοχή και ε, εντείνεται η ένταση μεταξύ Αρμενίας και Τιμπερτζάν με κίνδυνο ένοπλης ε, σύραξης. Ε, πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τους έξι εταίρους μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο σεβασμός ε, των βασικών κανόνων της δημοκρατίας και η επίλυση των ε, εδαφικών διενέξεων είναι απαραίτητα. Αναφέρομαι στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δέχεται να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο το οποίο διασφαλίζει την εδαφική αικαιρότητα όπως έχει ζητήσει και αυτό το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για τον Νότιο Κάφκασο. Και δεν μπορεί το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αγνοεί τις αρχές για το σεβασμό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τώρα λοιπόν ο κύριος Στογιάνοφ έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον Κάφκασο. Είναι πολύ σημαντικό η περιοχή αυτή να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο, γιατί μέχρι τώρα η περιοχή αυτή έχει διαιρεθεί σε δύο ομάδες κρατών. Αυτή τη στιγμή η Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν επιθυμούν από κοινού με την Τουρκία να απομονώσουν την τρίτη περιοχή που είναι, την τρίτη χώρα που είναι σε αυτή την περιοχή, την Αρμενία. Αυτό είναι απαράδεκτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμποδίσει αυτές τις εξελίξεις γιατί θα καταστρέψουν όλα αυτά που επιδιώκει η ανατολική εταιρική σχέση. Όσον αφορά την Ουκρανία και την περίπτωση Τιμοσέγκο και εγώ πιστεύω ότι η κυρία Τιμοσέγκο έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη κάτι το οποίο αμφισβητείται γιατί κρατείται για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Ουκρανοί ε, δεν πρέπει να δεχθούν ε, καμία ζημιά ε, στα δικαιώματά τους και δυστυχώς αυτή τους έβλαψε και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Κύριε Σάρους Βόλσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν συγκρίνω την Ολομέλεια εδώ στη συζήτηση για τον Νότο και τη συζήτηση για την Ανατολή, πώς να το πω, είμαι λιγότερο αισιόδοξο και λιγότερο χαρούμενος ε, από, ε, από τους προλαλήσαντες. Εγκρίνω την πολιτική σας κυρία Άστον και κύριε Φίλε. Όλα τα κείμενα είναι καλά και οι προθέσεις, αλλά τι γίνεται στην πράξη. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είναι αρνητική η εξέλιξη και η δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης και των γεγονότων στο Νότο. Απέτυχε να συμφωνήσει η Euronest ε, για, στη Σύνοδο Κορυφής και έχουμε και αρνητική δυναμική ε, στην Ανατολή μας γιατί υποχωρεί η δημοκρατία. Η δική μας πρόταση ποια είναι, η δική μας προσφορά. Ε, δημιουργεί ε, αρκετή πίεση για την πολιτική μας στις ε, ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Στο Νότο μας προσπέρασαν οι εξελίξεις και βρεθήκαμε προεκπλήξεις. Δεν θέλουμε να γίνουν τα ίδια στην Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε και άλλη καλή πρόταση γιατί θα δούμε στο Γερεβάν, στο Μίνσκ και στον για νέα πλατεία τα χρήματα. Έχω μια ερώτηση για την Ουκρανία που δεν μπορώ παρά να την κάνω. Εσείς κυρία Άστον και κύριε Επίτροπε αποκλείεται το γεγονός ότι ο Γιαννούκοβιτς παίζει διπλό παιχνίδι ε, δηλώνοντας ότι πηγαίνει προς την Ευρώπη και ταυτόχρονα σαμποτάρει ε, τη δημοκρατία με την υπόθεση Τιμοσέγκο. Μας εκβιάζει ότι θα γυρίσει προς τη Ρωσία και εκβιάζει και τη Ρωσία ότι θα έρθει μαζί μας αλλά είναι μια δοκιμή αυτή για την Ουκρανία. Μέχρι το τέλος της Πολωνικής Προεδρίας θα πρέπει να εγκρίνουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, αλλά να ανηθούμε να την επικυρώσουμε. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Uh, Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν τη διάσκεψη κορυφής. Ε, απ' την άλλη πλευρά, ο, το γεγονός ότι το 2009 ε, η αντίστοιχη ε, διάσκεψη έδωσε όθηση σε κάποια στοιχεία και έκτοτε πολλά έχουν επιτευχθεί, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και ότι θα καταφέρουμε τελικά να διαμορφώσουμε μια πολιτική η οποία ε, θα είναι στο ύψος της Ευρώπης. Ε, νομίζω ότι ε, δεν πρέπει να είμαστε και απεσιόδοξοι όσον αφορά την δυναμική γιατί βλέπουμε τα ίδια μου τα μάτια ότι πολλοί από τους ανατολικούς εταίρους βλέπουν την, το μέλλον τους μαζί μας, βλέπουν ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Μόνο που πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αξιοπιστία. Νομίζω Νομίζω ότι η αναθεώρηση ενδιάμεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας έδωσε μία νέα όθηση όσον αφορά την πολιτική προς την ανατολική εταιρική σχέση και νομίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να επιτύχουμε αποτελέσματα αλλά μονάχα με την προϋπόθεση ότι ο ένας θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες του άλλου και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να πω και στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό είναι και το μήνυμα άλλωστε το οποίο έχουμε πάρει από όλους τους εταίρους μας. Ε, ε, θα πρέπει να έχουμε κοινό στόχο να γίνουμε εδώ μια, μια περιφέρεια ε, ταξιδίου χωρίς ανάγκη θεώρησης, ε, χωρίς την ανάγκη για βίζα. Τέλος, η συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για όλες τις άλλες ε, χώρες ε, και νομίζω ότι όλη αυτή η αναφορά στις ελληνικές εποχές ε, νομίζω ότι είναι ακριβώς ένας λόγος παραπάνω για να τα αλλάξουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Και που τήρησατε και το χρόνο σας και τώρα Έχουμε ένα μπλε, μια μπλε κάρτα παρακαλώ. Συμφωνείτε να δεχτείτε αυτή την μπλε κάρτα. Ναι βεβαίως. Ναι, μια ερώτηση έχω, κύριε Βιγγένιν. και ύστερα από αυτά που ακούσαμε βέβαια και από τον κύριο Σαρουσβόλσκι. Για την ε, προσφορά αυτή της Euronest, τι γνώμη έχετε. Είναι αρκετά ελκυστική. Ποια είναι η εμπειρία σας. Θεωρείτε ότι ίσως μπορεί να εξασφαλίσετε ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Ευχαριστώ για την ερώτηση έτσι μου δίνετε και την ευκαιρία σε αυτό το σύντομο χρόνο που έχω στη μου να πω δύο λόγια για τη Euronest. Ξέρουμε βεβαίω ότι δεν είναι δυνατό να υιοθετηθεί η έκθεση ε, λόγω ίσονο σημασία διαφωνία σε ίσονο σημασία θέματα. Και λέω ίσονο σημασία γιατί έχουν πολλά άλλα συμφωνηθεί ήδη στο πλαίσιο τη Euronest, πολύ πιο σημαντικά. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο θα λάβουμε υπόψη για μελλοντικέ συνεδριάσει. Η εμπειρία μου όμω λέει ότι και οι πέντε χώρε έχουν ενδιαφέρον να ε, συνεχιστεί αυτή η συνεργασία μέσα από τη Euronest. Είναι μια ζώσα δομή και πιστεύω ότι όλοι θα επενδύσουν και στο μέλλον πολύ ενέργεια και δουλειά. Αυτή είναι η εμπειρία που έχω από την επίσκεψη στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν μετά την ε, ολομελέτη της Euronest πριν από δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βίζεν, τέλειος ο χρόνος σας και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πιοτρόφσκι. Σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η ανατολική γειτονία είναι μία από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. και στο τελικό έγγραφο της ε, Συνόδου ε, θα καταγραφούν ασφαλώς, θα έπρεπε μάλλον να καταγραφούν συγκεκριμένε ε, δηλώσεις και δεσμεύσεις ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση για Θεοδωριστή την άρση δηλαδή της υποχρέωσης και θα πρέπει να συζητηθεί με σοβαρότητα εάν οι ανατολικές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Έννοιας μπορεί να, μπορούν να έχουν μια επιπλέον στήριξη όπως η περιφέρεια του Λιούμπλιν στην ε, Πολωνία θα μπορούσε να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Στην ε, πολιτική γειτονία υπάρχουν ε, αντίστοιχα παραδείγματα σε σχέση και με τον δυτικό χώρο αλλά και με τον ανατολικό. Δεν θα πρέπει τα πολιτικά προβλήματα που γνωρίζει η Ουκρανία να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη αυτής της εταιρικής σχέσης το σενάριο της, της ε, Αραβικής Άνοιξης ε, καλύτερα να μην επαναληφθεί. Εάν δεν διατεθούν τα χρήματα την ώρα που πρέπει, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουγγουριάνο, 1,5 λεπτό. αναγνωρίστηκαν οι φιλοδοξίες των ανατολικών μας εταίρων από την τελευταία ε, διάσκεψη Euronest. Αρκεί αυτό όμως. Και τι θα γίνει με τις πολιτικές ε, πραγματικότητες που βλέπουμε να αναπτύσσονται στα ανατολικά μας σύνορα όταν η Τιμοσέγκο ε, υπόκειται σε μια σταλινιστικού τύπου δίκη. Θα πρέπει πιστεύω να επανεπιβεβαιωθεί η δημοκρατική εναλλακτική λύση κατά της μετάδοσης της, ε, του καθεστώτος Πούτιν και σε άλλες χώρες. Βέβαια τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι πιστικά. Η απελευθέρωση του καθεστώτος ε, ίσων διαβατηρίου προχωρά αλλά με, αργά, ε, με αργή, αργό ρυθμό. Υπάρχει απογοήτευση και οι εταίροι μας ε, θεωρούν ότι έχουν υποβαθμιστεί οι νότιοι σε σχέση με τους ανατολικούς. Ε, ούτε και στον Αμπούκο φαίνεται να υπάρχει απαιτουμένη πρόοδος. Ε, η δυνατότητα μετριασμού της Ένωσης μπορεί να βοηθήσει στις περιπτώσεις που έχουν αυτά τι λεγόμενες παγωμένες συγκρούσεις. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κάτι καινούριο στο ανατολικό μέτωπο Υπάρχει έλλειμμα πολιτικής βούλησης ε, και αυτό δεν ε, ενθαρρύνει τους εταίρους μας να προβούν σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και αυτό θα μπορούσε να προσθέσει μια στρατηγική και ενεργειακή κρίση η οποία θα πολλαπλασιάσει την οικονομική κρίση που ήδη γνωρίζουμε. Η ανατολική διάσταση των πολιτικών μας είναι μια πολιτική πρέπει να την αναπτύξουμε εμείς. Διακόπτεται ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ. sorry. We have to continue. Λυπούμε, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε με την κυρία Φλασικόβα που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητή κυρία είπατε πρόσωπε, καταλαβαίνουμε ότι τους τελευταίους καιρούς ε, έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στα νότια σύνορα της Ένωσης σχέση με τα ανατολικά. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους ανατολικούς μας εταίρους μετά την ε, διεύρυνση του 2004 έχουμε δημιουργήσει μια νέα γειτονική σχέση, μια μεγαλύτερη γειτονιά και για αυτές τις χώρες θα πρέπει να δώσουμε νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες. Η δυνατότητα της συνάντησης της Βαρσοβίας ε, δεν θα πρέπει να παραμεληθεί. Το 2011 ε, θεωρείται κρίσιμο και πολύ σημαντικό για το μέλλον και ένας ε, πολύ σημαντικός τομέας είναι η χρηματοδότηση. Παρά τις προσπάθειες του 8 και του 2013 θα έχουμε αύξηση με το χρηματοοικονομικών πόρων, αλλά έχουμε την πρόκληση για τη μελλοντική δημοσιονομική περίοδο. Να δούμε τι θα γίνει εκεί με την αύξηση της χρηματοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ρωσίας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα έξι μέλη της Προσωπητικής Ένωσης. Η εταιρική σχέση δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως μια δραστηριότητα κατά της Ρωσίας. Ε, τέλει θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι με τέτοια πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να αφήσει να χαθούν οι καλές ε, ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν με την Πολωνική Προεδρία και θα πρέπει να αναβαθμίζεται αυτή η πρωτοβουλία συνεχώς με τη συμμετοχή όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, στη δεκαετία του 90 Θυμάμαι πολύ καλά πώς άρχισε να εκδηλώνεται η προοπτική για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Πολωνία. Πράγμα το οποίο μας βοήθησε όλους να αναπτύξουμε και να διαφυλάξουμε δημοκρατικές ε, αρχές και προδιαγραφές. Οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουν ε, να προωθήσουν ε, νέες αρχές από ό,τι βλέπω και αξίες. Έχουν παρατείνει την εποχή του λίθου κατά τέσσερα χρόνια. Πρέπει νομίζω να απευθύνουμε έκκληση σαφή μέσα από την διάσκεψη της Βαρσοβίας, όπως είπε και ο κύριος Σίλιτς, για μια ε, προοπτική για τις χώρες αυτές, προοπτική που θα τις βοηθήσει στη γεωπολιτική τους κατάσταση, προοπτική που θα τις βοηθήσει τι χώρε αυτέ να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό Πρόεδρε θα ήθελα να αποσταλεί ένα σαφέστατο μήνυμα από τη Βαρσοφία, ένα, σύστημα, ένα μήνυμα ενσωμάτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γκάλερ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, η Ανατολική γειτονία έχει μεγάλη σημασία και για μας και για του εταίρου μα στα Ανατολικά σύνορα δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Το more for more είναι η, προσέγγιση που έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερα για περισσότερα, αντί για το λιγότερα από... για λιγότερα, less for less, που βλέπουμε μερικέ φορέ να εφαρμόζεται. Για την Ουκρανία βλέπω ότι έχουν συμφωνήσει στη Γιάλτα τα τρία θεσμικά όργανα την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, με τον κύριο Μπροκ, με τον κύριο Φίλε για μία πρόοδο που θα άφηνε πίσω της την περίοδο του ε, σταλινισμού. Ο, ο Γιακούνοβιτς θα πρέπει να δεχθεί το κράτος δικαίου, θα πρέπει να προσμετρηθεί η αξία του με βάση τα δεδομένα και τα κριτήρια του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. προσπαθούν κάποιοι να αναπτύξουν ε, μια επιτροπή για, την, ε, για το τέλος του σταλινισμού, για την επάνωση στη δημοκρατία, γιατί πιστεύουν ότι έτσι μπορεί να βοηθήσουν τη χώρα τους. Αντιλαμβάνομαι τις επικρίσεις που ακούστηκαν από συνάδελφο για την κατάσταση της δημοκρατίας και στη Ρωσία, για την εκλογική αναμέτρηση που ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να αποστείλουμε παρατηρητές, γιατί είναι δεδομένο ήδη ότι δεν θα είναι δίκαιες και ανώθευτες οι εκλογές. Αυτές λοιπόν οι επικρίσεις ε, κατά της Ουκρανίας που ακούγονται σήμερα θα πρέπει να διατυπώνονται εφραδός και ευθαρσός και κατά ενός μεγαλύτερου ακόμη εταίρου μας της Ρωσίας. Ευχαριστώ πολύ. Είστε διατεθειμένος να δώσετε απάντηση σε μια μπλε κάρτα. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα επακριβώς αυτό που είπατε στο τέλος της παρέμβασής σας. Δεν θέλετε να αποστείλουμε αντιπροσωπεία παρατηρητών στη, στα κράτη εκείνα στα οποία υπάρχουν υπόνοιες για ανώθευση των εκλογών. Δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο σας κινεί σε αυτή την τοποθέτηση. Διότι οι παρατηρητές ε, ε, θα μας ενημερώσουν για προβλήματα, παρατυπίες, ε, ε, νοθεί ενδεχομένω. Θα πρέπει ακόμη και αν έχουμε την υπόνοια ότι θα είναι νοθευμένε οι εκλογέ να αποστείλουμε παρατηρητέ στη Ρωσία. Κύριο Σκάλερ. Ε, εγώ που είμαι και επικεφαλή παρατηρητής των εκλογών για την Τινησία πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει οι αποστολές αυτές παρατηρητών να γίνονται μόνο εκεί όπου είμαστε πεπισμένοι ότι η διαδικασία μπορεί εν όλο να οδηγήσει σε ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα. δυνάμια έστω. Και δυστυχώς, δυστυχώς βλέπω ότι στη Ρωσία και δεδομένων και των πρόσφατων εξελίξεων, είναι δεδομένο ότι αυτή η διαδικασία δεν πρόκειται να οδηγήσει σε μια ε, δίκαιη εκλογική αναμέτρηση και εκλογική διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι οργανωμένο και δομημένο όλο το όλος ο μηχανισμός ε, στη Ρωσία, ο εκλογικός μηχανισμός και οι διαδικασίες που να ε, επιτρέπουν την απονομή του τίτλου δίκαιε και ανώθευτε εκλογέ στη Ρωσία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνο να προσφέρουμε παρατηρητέ. Ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Πάσκο παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ανατολική εταιρική σχέση είναι η απάντηση ε, και η εναλλακτική ε, λύση όσον αφορά ε, την ενέργεια και όσον αφορά τους αγωγούς ενέργειας. Αυτές οι χώρες είναι χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής της Τέος Ενώσεως και επομένως πολλά πράγματα θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή. Η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί με την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το νέο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής δημιουργεί οπωσδήποτε περισσότερα προβλήματα και δυσχεραίνει την κατάσταση, δυσχερεί από την οποία προσπαθεί να ωφεληθεί η Ρωσία. Όμως οι συμφωνίες σύνδεσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να μην αλλάξουν τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Μιέλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Σύνοδος Κορυφής για την Ανατολική Γειτονία έχει ασφαλώς για την Πολωνία τη σημασία του μεγαλύτερου γεγονότος που την αφορά. Η δήλωση μπορεί να αποτελέσει μια, ένα πολύ καλό έγγραφο για την συνεργασία της, των Βρυξελών με, την, ε, με τους γειτονές, τους, ε, τους γειτονές μας προς τα ανατολικά. Είναι πολύ μεγάλη σημασία των κρατών αυτών και ενισχύεται διαρκώς. Γι' αυτό όλο και περισσότεροι από τη δική μας πλευρά ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη καλών σχέσεων ανατολική γειτονία. Τέτοια έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν καλή βάση, πιστεύω, και, πιστε... και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορέσουμε να υπογράψουμε μια συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία ε, όπως άλλωστε έχουμε την ευκαιρία και με τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, η οποία θα βοηθήσει τα μάλλα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, οι σχέσει, η βελτίωση των σχέσεων με την ε, Γεωργία και τη Μολδαβία αποτελούν ένα ε, πολύ θετικό ε, βήμα. Και η κοινή διοργάνωση και συνεργασία μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας το 2012 πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Τα ευρωπαϊκά κράτη λοιπόν θα πρέπει σε όλε αυτέ τι εξελίξει που διαπιστώνουμε στα ανατολικά μα σύνορα να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Ήμπρι για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στα ανατολικά μας ε, σύνορα ε, αυτή τη στιγμή έχουν, ε, βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, έχουν ξεκινήσει την διαδικασία εκδημοκρατισμού. Είναι μεγάλη η πίεση της κοινωνίας των πολιτών, αλλά χωρίς ειρήνη και σταθερότητα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πολλοί συνάδελφοι που μίλησαν μέχρι τώρα αναφέρθηκαν στον Αγκόρνη Καραμπάχ και ε, αυτά τα οποία συνέβησαν, οι εντάσεις οι οποίες συνέβησαν την άνοιξη εκεί. Και βεβαίως κατεδείχθη ότι όταν ε, συνεργαζόμαστε εμείς ε, τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Ήταν σαφές αυτό κυρία Άστον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει τίποτα να κάνουμε άλλο σε αυτή την περιοχή. Αντιθέτως, δεν πρέπει καθόλου να εφηζηγάζουμε. Θα πρέπει και η κυρία Άστον πιο συχνά να μας εξηγεί τι συμβαίνει ε, σε αυτές τις παγωμένες ε, διαμάχες. Επίσης, δεν υπάρχει μονάχα τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ε, υπάρχει και η Περνιστερία, υπάρχουν και άλλες ε, περιοχές και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να αντιμετωπίζει όλες αυτές ε, τις περιοχές τριβής και βεβαίως και οι δράσεις και τα έργα θα πρέπει να διαφέρουν αναπερίπτωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυρίλοφ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, προσφέρει πολλέ ευκαιρίες για αποδοτική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανατολικών Εταίρων ε, η Ανατολική Εταιρική Σχέση. Πιο σημαντικό όμω είναι αυτή η προσθέμενη αξία που προσφέρει η πολυμερής διάσταση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, επικεντρώσουμε σε ξεχωριστέ χώρες, αλλά να αναπτύξουμε το δυναμικό όλης της γειτονικής αυτής περιοχής, να διατηρήσουμε την ισορροπία δηλαδή στη σχέση με όλες τις χώρες. Περιφερική περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική, ιδίω η ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, διάδρομη σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης, αλλά και σημαντικό στοιχείο της οικονομικής ολοκληρωσής ε, των εταίρων μας στην Ένωση. Δυστυχώς είναι ε, αδύνατο να υπάρξει συνεργασία όταν υπάρχουν συγκρούσεις και κλειστά σύνορα. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνη και ειρήνη και να κλιμακώσουμε τι προσπάθειέ μα για την εξέβρεση μια ειρηνική λύση ε, στι ε, ανεπίλητε συγκρούσει περιοχή. Ε, είναι σταθεροποιητικό ο Ρώσο Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γεωργία, αλλά θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε ό,τι αφορά την υπερδημιστερία και τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στα θέματα αυτά και στο πλαίσιο του διαλόγου Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσίας που είναι πολύ σημαντικό. Σαφεί δεσμεύσει είναι επίση απαραίτητε από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση για την συμμετοχή μετά την σύγκρουση και για την σταθεροποίηση. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την ανατολική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κόβαλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, δεν συμμερίζομαι την έποψη ότι, έχουν γίνει, ότι, ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για την Ανατολική Γειτονία. Φαίνεται μάλλον ότι η Ευρώπη ε, ε, την έχει βάλει στο περιθώριο, εκτός από τα εμπορικά θέματα. και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά αυτή την ε, στράτευση στην υπόθεση Ανατολική Γειτονία. Εγώ παρακολούθησα εκ του σύνεγγυ τη εργασίε τη Συνόδου Κορυφή τη Βαρσοβία και πρέπει να γνωρίσουμε τι σημαίνει αυτή η Σύνοδο Κορυφή. Θα πρέπει. Εγώ θα παρακολουθήσω μάλλον ε, και έχω μέχρι τώρα παρακολουθήσει προσεκτικά τι εξελίξει αυτή τη Σύνοδο Κορυφή και θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει δηλαδή όταν έχουμε μια γενιά ανθρώπων νέων που μεγαλώνουν πάνω στο σχολείο, τελειώνουν και. θα είναι η γενιά με την οποία θα συναλλαγόμαστε εμείς. Χρειάζεται δηλαδή ένα πανεπιστήμιο το οποίο να προετοιμάσει τη γενιά αυτή, μια γενιά μια νέων παιδιών, στην, ε, για μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και προοπτικές βέβαια γενικότερα για την ε, Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κουσίπ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Ήταν πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που απέστειλε η Πατή εκπρόσωπος. Μιλήσατε για πολύ καλά αποτελέσματα της ε, Ανατολικής Γειτονίας. Σας το εύχομαι και σας και στον κύριο Φιούλε και στην Πολωνική Προεδρία. Βέβαια θα ήθελα να μην ε, χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα όπως ε, είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε στο στη συνέχεια της συνόδου της Euronest. Θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα από τις συνοδοκορυφές της Βαρσοβίας. Και τι εννοώ με αυτό. Εγώ περιμένω μια ενιαία διαμόρφωση, μια ενιαία θέση για την χρηματοδότηση της Ανατολικής Γειτονίας. Αναμένω να γίνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να στηριχθεί η αντιπολίτευση στην ε, Ουκρανία, η αντικοθεστατική όπως η κυρία Τιμοσέγκο. Θα πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις πιο στενές με τη Μολδαβία και τη Γεωργία και πρέπει πιστεύω να ανοίξουμε τις πόρτες μας και προς την Λευκορωσία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της ε, Ανατολικής Γειτονίας όλοι μεταξύ μας με κίνητρα. Κίνητρα Φερρυπίν όπως η άρση της υποχρέωσης θεωρής διαβατηρίου. Δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση για τους υπηκόους ε, της Ρωσίας. Αλλά ε, το Σέγγεν φραγμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ορθώνεται μπροστά στα κράτη της Ανατολικής Γειτονίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την Ουκρανία και για τη Μολδαβία και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης χρειάζεται στήριξη για την ανάπτυξη υποδομών, ιδιαίτερα και στην κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η δεύτερη σύνοδος κορυφής της εταιρική σχέση στη Βαρσοβία είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να δοθεί ένα πιο ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας καθώς τα συμπεράσματα της συνόδου θα έχουν ουσιαστική σημασία στη μελλοντική εφαρμογή της ανατολικής εταιρικής σχέσης. οπωσδήποτε πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική γειτονίας και βέβαια το κείμενο της ευρωπαϊκής επιτροπής μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει είναι και σημαντικό και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. ωστόσο υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν έχουν γίνει τα βήματα που πρέπει υπάρχει αποσπασματικός τρόπος με τον οποίο έχει προχωρήσει η πολιτική γειτονίας και όχι πάντα με ευθύνη δική μας. βεβαίως η δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παραμείνει πάρα πολύ ισχυρή από δικής μας πλευράς και ταυτόχρονα η στήριξη πρέπει να παρέχεται υπό όρους και να εξαρτάται από την πρόοδο που γίνεται από την κάθε χώρα χωριστά. ουσιώδους σημασίας βέβαια είναι και η προσέγγιση προς την κοινωνία των πολιτών και αποτελεί θετική εξέλιξη τέλος η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για τη δημοκρατία σαφέστατα είναι ευπρόσδεκτη και απευθύνομαι και στην ύπατη εκπρόσωπο και στον επίτροπο όμως αυτό θα καθυστερήσει για να δημιουργηθεί και ταυτόχρονα έχουν μείνει κονδύλια και εργαλεία τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως πρέπει. έχουν αξιοποιηθεί μερικώς και νομίζω ότι εκεί πρέπει όσο ότου δημιουργηθεί αυτό το ευρωπαϊκό ταμείο να πέσει το βάρος της Ευρωπαϊκή επιτροπής βέβαια με την ε, αποφασιστική σημασία πολιτική απόφαση του συμβουλίου που είμαι βέβαιη πως θα εξέλθει από τη σύνοδο της βαρσοβίας. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή αλλαγή τώρα στη σειρά των ομιλητών. Ο κύριος Κούκαν πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η διάσκεψη κορυφή Βαρσοβία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη Πολωνική Προεδρία και πιστεύω ότι θα αποτελέσει σταθμό στι σχέσει μα με του ανατολικού μα εταίρου όταν η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στην εξωτερική της πολιτική. Πρέπει να βρούμε στρατηγικούς σημαντικούς εταίρους. Πρέπει να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε ένα μείζωνα ρόλο στην περιοχή αυτή. Αν θέλουμε να πετύχει τώρα όμω η ανατολική εταιρική σχέση, πρέπει να καταστεί πολιτική εταιρική σχέση. Θα πρέπει να εντείνουμε τι σχέσει μα. Θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίε και να υιοθετήσουμε ένα όραμα που θα εμβαθύνει την συνεργασία των χωρών αυτών με την Ένωση. Η διάσκεψη κορυφή αυτή λοιπόν είναι η ευκαιρία μα να ορίσουμε την ατζέντα, του στόχου μα για την επερχόμενη περίοδο που ίσω να είναι και αποφασιστική σημασία. Διαφορετικά αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι οι χώρες αυτές θα δράσουν καιροσκοπικά, οπορτουνιστικά και ίσως τα πράγματα παγώσουν κάπου μεταξύ του σοβιετικού παρελθόντος και της δημοκρατικής μεταρρύθμισης. Αυτό δεν θα ήταν προς όφελός μας, εξού και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε ζητήματα όπως είναι απελευθέρωση καθεστώτος θεωρήσεων, ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών. Και κάτι τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα ζητήματα της ασφάλεια και των εμπορικών σχέσεων, ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερο τι χώρε αυτές και να τους δώσουμε τη δυνατότητα και αυτοί να μας προσεγγίσουν. Και ελπίζω να στεφθεί εύχομαι με επιτυχία διάσκεψη κορυφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μικολάσικ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Σύνοδος της Βαρσοβίας δίνει ελπίδα και μάλιστα ελπίδα αναβίωσης ε, στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τους ανατολικούς γειτόνους. Χρειαζόμαστε όμως μια ε, νέα στρατηγική έτσι ώστε να επιτευχθούν αμεσότερα οι στόχοι. Η ανατολική εταιρική σχέση μπορεί να αποτελέσει ένα καλό όχημα αμοιβαίας εποφελούς σχέσεις και βεβαίω πάντα μέσα στα πλαίσια του σεβασμού των υποχρεώσεών μα. Ε, πιο ε, σαφής γραμμέ θα πρέπει να καθορίσει η διάσκεψη της ε, Βαρσοβίας και όσον αφορά χώρε όπως η Ουκρανία θα πρέπει οπωσδήποτε ε, στις γειτονικές μας χώρες να βοηθήσουμε την ενδυνάμωση και εμβάθυνση της ε, δημοκρατίας χωρίς να ξεχνούμε ε, τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται η πρώην Πρωθυπουργός Τιμοσέγκο. Ε, όταν ε, αναφερόμαστε σε εξελίξεις δεν μιλάμε μόνο για την οικονομία αλλά ε, και για την ενέργεια και την ασφάλεια και βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα και ε, ε, μην ξεχνούμε και διάφορες ε, περιοχές όπου οι τριβές εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Επίσης δεν πρέπει να αγνοούμε κάποιες υποχρεώσεις από πλευράς της Αρμενίας που στηρίζει η Ρωσία. Θα πρέπει να βρούμε συνολικά μια νέα προσέγγιση. Είναι ο κύριος Τόκες. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, η διάσκεψη κορυφή Ανατολική Εταιρική Σχέση στη Βαρσοβία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο όπως και επί Ουγγρικής Προεδρίας και επί Πολωνικής Προεδρίας είναι πολύ σημαντικό θέμα στην ε, ατζέντα. Και αυτές οι χώρες είναι και σημαντικοί εταίροι ε, στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής της Συνόδου Κορυφής. Και θέλω να επενέσω βέβαια και τις χώρες αυτές αλλά και τη Σουηδία που ήταν κινητήρο μοχλό τη ε, της προετοιμασίας. Θα ήθελα να πω ότι και εμείς που είμαστε πριν στο Σοβιτικό Μπλοκ, ε, η Ουγγρική Αλληλεγγύη έχει δείξει μεγάλη αλληλεγγύη και στην πανταξιακή διαδικασία της Κροατίας. Η Πολωνία τώρα δείχνει το δρόμο στην Ουκρανία. Στην 20η επέτειο της ε, πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης είναι πεποίθησή μου βαθιά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαιρέθηκε τα μάλλα, μπορεί να επανενωθεί και με την άλλη πλευρά του σιδηρού, σιδηρού παραπετάσματος αλλά μόνο εάν εφαρμοστούν σωστά οι διαδικασίες ολοκληρώσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι έγινε στη γειτονιά μας ε, και αν ε, ό,τι γίνεται επηρεάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και η σωστή πολιτική από πλευρά Ένωση. Οι χώρε ε, τη Ανατολική Εταιρική Σχέση πραγματοποιούν μεταρρυθμίσει για να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχώ ζητούμε από τι χώρε αυτέ περαιτέρω μεταρρυθμίσει. Την ανάγκη να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα, παραδείγματο χάρη στη Λευκορωσία, στην Ουκρανία. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι στη δέσμευσή μα, να θεσπίσουμε στενότερου δεσμού και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάσκεψη κορυφή για να στείλουμε το σωστό πολιτικό μήνυμα τη πολιτική βούληση που έχουμε να παίξουμε έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Θα περάσουμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε λάβει, το Προεδρείο έχει λάβει πολλά αιτήματα, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όλα, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας πέντε λεπτά. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Λίσεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπατή κύριε Επίτροπε, ως Πολωνός αισθάνομαι περήφανο που μπορούμε Εμεί να έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τη Σύνοδο Κορυφή ε, στην Πολωνία. Και Μπορεί να είναι υπερήφανη όχι μόνο η Πολωνία αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει νέα προοπτική και εξελίξει σε αυτά τα έξι κράτη τα οποία περιμένουν να δούνε το πρόγραμμα ε, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, αλλά και που θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση, στην πολιτική, τη δημοκρατία, την ασφάλεια. Θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες και δίνεται η εντύπωση ότι θα ήταν πολύ θετικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Είναι πολύ θετικό το να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τη συμφωνία σύνδεσης ε, με την Ουκρανία αλλά και με την ε, Μολδαβία και τη Γεωργία.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 Η ανατολική εταιρική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική για, τη, για έξι χώρες Ανατολικής Ευρώπης ε, και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως τα αποτελέσματα δεν θα είναι άμεσα. Θα τα δούμε σε μερικά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της πολιτικής την χείρα βοηθείας προς τις χώρες αυτές. της οδηγεί ε, στην οδό της δημοκρατίας και στην βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου. Σήμερα μιλήσαμε το πρωί για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη και επομένως θα πρέπει και προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την περιοχή μάλλον τη γεωγραφική να ενδυναμώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις, ε, να υπάρχει αμοιβαία ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου. κεφαλαίου. Η βελτίωση της οικονομικής ε, ζωής ε, θα ε, διευκολυνθεί και από την άρση της ανάγκης βίζας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Thank you very much. Parteneriatul Estic reprezintă o oportunitate deosebită pentru Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Ανατολική Γειτονία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα κράτη της Ανατολικής Γειτονίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οικονομική και την πολιτική τους σταθεροποίηση, για την ευημερία τους. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2009 θα πρέπει να συνεχιστεί και να εδραιωθεί. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για το γεγονό ότι η Προεδρία τη Πολωνία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στην, στην ε, πτυχή αυτή και περιμένουμε να δούμε και τα συμπεράσματα τα σχετικά με την πορεία της υλοποίησης ε, των μέτρων και των προτάσεων. Επίσης, τα μέτρα που θα αναλυφθούν θα πρέπει να στοχεύουν πριν τους πολίτες έτσι ώστε και αυτοί να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, δημοκρατία, ευημερία. Θα πρέπει όμως ε, να διαθέσουμε και τα απαιτούμενα κονδύλια για αυτή την προσπάθεια στην περίοδο 2014-2020 προς το χρηματοδότηση δηλαδή. Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η διάσκεψη κορυφής της Βαρσοβίας πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πρώην Σοβιετικών ε, κρατών. Θα πρέπει να δοθεί νέα όθηση. Για του εκπροσώπου τη Ανατολική Εταιρική Σχέση, η Βαρσοβία θα είναι παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί με τη δημοκρατική αλλαγή σε μια χώρα που ήταν ε, πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι έχουν τη δική τους δημοκρατία, έχουν βέβαια ελλείμματα σε τη διαχείριση της χώρας τους και θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι πρέπει να προσέξουν τους πολίτες τους και θα πρέπει η Βαρσοβία να τους στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Πρέπει να ζουν ε, σε ειρήνη και δημοκρατία. Και πρέπει βέβαια να προσέξουμε αυτές τις ηγεσίες γιατί είναι αυτοί που εκπροσωπούν πολιτικά ε, τους πολίτες των χώρων. Κυρία Μορβάη παρακαλώ. Κυρία Μορβάη, Πρόεδρε, μουσική στα αυτιά μου συζήτηση για το σταλινισμό και τη μεταρρύθμιση εδώ στην Ολομέλεια. Όμως είναι λίγο παρά, ε, παράτονη αυτή η μουσική, διότι ακούγονται και αντίθετες απόψεις. Θα πρέπει να θυμίσω ότι η Judith Τσίμερ είναι μια συνδικαλίστρια στην Ουγγαρία, η οποία οργάνωσε συλλαλητήριο, συνελήφθη βρίσκεται εδώ και μήνες στις, ε, στο κρατητήριο. Στη Θεοκαρία δύο αντικαθεστατικοί, δύο μέλη της αντιπολίτευσης βρίσκονται και αυτοί στη φυλακή. Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες προχωρούν ενώπιον των δικαστηρίων και κλεισμένων των θυρών, όπως και ο οποίος δεν είναι, ε, ο οποίος βρίσκεται ε, στο εδόλιο του, ε, ε, κατηγορουμένου, αλλά χωρίς να δυνατέ να παρίσταται στην ίδια του τη δίκη. Αυτά είναι η εποχή του στελινισμού, η οποία συνεχίζεται και στην Ουγγαρία ακόμα. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Ο είναι ο τελευταίος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, αρκετά κράτη-μέλη τα οποία τάσσονται ε, στέκονται μάλλον επιφυλακτικά έναντι της Λευκορωσίας και του καθεστώτος της και έναντι της ε, Ουκρανίας επίσης. Πιστεύω όμως ότι η πολωνική Προεδρία επεξεργάζεται τα θέματα αυτά κατά τρόπο ε, συνεπή και προσεκτικό και θα πρέπει να συνεχίσει να διατηρήσει αυτή την ε, προσεκτική και συνετή στάση στις σχέσεις με τα κράτη της Ανατολικής Γειτονίας. Θα πρέπει να δώσουμε νέα όθηση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών Ανατολικής Γειτονίας και θα ήθελα να αναφερθώ και στην ενσωμάτωση η οποία θα μπορούσε να περάσει και μέσα από την ε, Επιτροπή των Περιφερειών, παραδείγματι. Στο Μπούζενστατ είχαμε, είχαμε τέτοιε εκδηλώσει, παραδείγματι, σε 7 Σεπτεμβρίου. Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλεια, την Κάθριν Άστον, να πάρει το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ πολύ, κυρία ε, Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Οι εξωτερικοί βουλευτές έθιξαν ε, πολλά ζητήματα και θα ξεκινήσω ε, με, ε, τον λόγο, με την ερώτηση γιατί κάθομαι σε αυτή την πλευρά και όχι στην άλλη. Κοιτάξτε, το ίδιο πράγμα θα ήταν και στη μέση να καθόμουν, πάλι ευτυχής θα ήμουνα. Το ζήτημα είναι να αντιμετωπίζουμε σωστά τα πράγματα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ερώτημα το οποίο τέθη ε, ε, στην ε, συζήτηση αυτή είναι εάν και κατά πόσον έχουμε την πολιτική βούληση έτσι ώστε να προωθήσουμε την ανατολική εταιρική σχέση έτσι ώστε να δούμε πραγματικά τις ανάγκες των γειτόνων μας. Και εγώ είπα, αλλά και πολλοί από τους παρεμβαίνοντες ε, και πολλοί από τους παρεμβαίνοντες ε, ανέφεραν ε, πράγματα τα οποία είναι σαφή και νομίζω ότι εξ αυτών συμπεραίνουμε ότι η απάντηση είναι θετική. Ναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πολωνική Προεδρία για την τρομερή εργασία, την πολλή δουλειά που έχουν κάνει και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες των οποίων δεν έχουν φυστεί μέχρι τώρα έτσι ώστε να να ε, οργανωθεί η Σύνοδος Κορυφής και ώστε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεω η αντιπροσώπευση να είναι ε, σωστή. Δεν υποτιμώ ε, τα διακυβεύματα τα οποία σχετίζονται με τους έξι εταίρους μας. Ο καθένας από τους εταίρους αυτούς, η κάθε μία από τις χώρες αυτές, φέρνει μαζί της μία πρόκληση, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έγινε λόγο σήμερα πολλής ε, και ε, για τις ε, διαμάχες οι οποίες είναι παγωμένες και για ενδεχόμενα νέα πεδία διαμαχών τα οποία θα προκύψουν, για προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα ανακύψουν. Όμως το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με τρόπο σαφή και διάφανο. Νομίζω ότι ε, ένα άλλο θέμα το οποίο συχνά αναφέρθηκε στη συζήτησή μας είναι το θέμα της Ιουλίας Τιμοσένκο. οι επικρίσεις ε, όσον αφορά αυτήν την κατάχρηση του δικαστικού συστήματος ε, δεν προέρχονται μονάχα από μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θίξει και εγώ απέναντί τους και ο Στέφαν επίσης. Νομίζω ότι αυτές ε, οι δικαστικές διαδικασίες πρέπει να είναι σωστές. Αυτό θέλουμε εμείς. Θέλουμε ένα σωστό δικαστικό σύστημα. Θέλουμε ανθρώπους τους οποίους το δικαστικό σύστημα ε, θα τους φέρεται με τρόπο ορθό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το ε, ε, ζήτημα ε, στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τις χώρες αυτές και δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει αυτές τις βασικές αξίες και αρχές της. Πιστεύουμε πάντως ότι η ανατολική ετορική ε, σχέση ε, πρέπει να προχωρήσει γιατί ακριβώς ε, παρέχει τα εχέγγυα για διευθέτηση τέτοιων προβλημάτων και όταν τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν επικυρώσει τις ειδικέ συμφωνίες τότε ο δρόμος θα είναι πιο εύκολος. Ε, όσον αφορά το εργαλείο για την πολιτική γειτονία, έχουμε ήδη ε, ορίσει 22 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά αυτό το χρηματοδοτικό ε, εργαλείο, το οποίο βεβαίως θα το διαχειριστούμε με τρόπο ανοιχτό και διαυγή αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να υπάρχουν επικαλύψεις με εργαλεία τα οποία έχουμε ήδη, αλλά να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και να προσπαθήσουμε να τα ε, στηρίξουμε. Ε, ε, θα πρέπει να βρούμε δηλαδή τρόπους για να στηρίξουμε πιο αποτελεσματικά τον, τον κόσμο, του, τους πολίτες των χωρών αυτών, τις πολιτικές εξελίξεις και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε πραγματικά μια προστιθέμενη αξία απέναντι στους ανθρώπους που χρήζουν σας. Θα τελειώσω εστιάζοντας για μία ακόμα ε, φορά ε, στα αναμενόμενα από την Σύνοδο Κορυδής αυτής από την μία πλευρά έχουμε ε, την συμφωνία με την Ουκρανία και την, τον χώρο ελεύθερων συναλλαγών. Επίσης, ε, εγώ ε, θα ήθελα να προχωρήσει το θέμα της Μολδαβίας. Το ζήτημα της κινητικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε σύντομα. Όσον αφορά τώρα την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων, κυρίως δε όσον αφορά τις μεταφορές, βεβαίως είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά και πάνω απ' όλα η πολιτική βούληση αλλά και η συνέχιση του πολιτικού διαλόγου θέλουμε να συνεχίσουμε ε, την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με τους ε, ανατολικούς ε, εταίρους. Να έχουμε δεσμεύσεις οι οποίες θα είναι σημαντικές αλλά και να λογοδοτούμε για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε. Πιστεύω ότι θα δοθεί νέα όθηση και νέα ενέργεια στην εργασία μας μέσω αυτής της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ε, και η ε, Ουγγρική Προεδρία έκανε ε, πολλή δουλειά και είμαι βεβαία ότι στη Βαρσοβία τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια πολύ σημαντική σύνοδο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα προχωρήσουμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, δύο λεπτών, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που αφορά στον γενετήσιο προσανατολισμό και στην ταυτότητα του φύλου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω να επιστρέψετε στις θέσεις σας. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας,